Uh, Κυρίες και κύριοι, να σας καλέσω να καθίσετε και να σας καλωσορίσω στην ε, δεύτερη μέρα της συνεδρίασής μας. Η σημερινή συνεδρίαση, όπως συνηθίζεται πια με τις συνεδριάσεις μας, ε, μεταδίδεται μέσω διαδικτύου να καλωσορίσω λοιπόν και όποιον ξύπνησε αρκετά νωρίς ώστε να μας ακούσει. Και Να σας θυμίσω ότι στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε την μηνιαία εφημερίδα μας και αυτόν το μήνα ειδικά μπορείτε να δείτε και το σχέδιο εργασίας της Επιτροπής μας για το 2011. Βρίσκεται και αυτό στην ιστοσελίδα μας. Ε, σας καλώ λοιπόν να το καλέσετε και μπορείτε επίσης να γίνετε φίλοι εντό εισαγωγικών με την Επιτροπή μας. Χωρίς μικρόφωνο μιλητής. Sorry, the microphone Ζητώ συγγνώμη, έσβησε το μικρόφωνο. Ελπίζω να ακούσατε το διαφημιστικό μου μήνυμα. Όπως και να έχει, είναι ιδιαίτερη χαρά σήμερα να καλωσορίσω σήμερα στη συνεδρίασή μας τον Ζόλταν Σέφερβεϊ που είναι ο ε, Ούγγρος ε, Υπουργός Οικονομικών και ε, ασχολείται με θέματα εσωτερικής αγοράς, ε, είναι φανατικός οπαδός της εσωτερικής αγοράς το φθινόπωρο είχα τη χαρά να διπνήσω μαζί του στη Βουδαπέστη, όπου είχαμε μια πολύ ζωντανή συζήτηση για κάποια από τα θέματα που ε, μας απασχολούν και ιδιαίτερα την, ε, ε, την νομική πράξη για την ενιαία αγορά. Χαίρομαι λοιπόν που είχατε την ευκαιρία να έρθετε στην Επιτροπή μας στην αρχή της Προεδρίας σας. Ξέρω ότι θα μα μιλήσετε και για το θέμα αυτό και για άλλα που σας ενδιαφέρουν. Ε, κυρίως όμως ε, σας καλωσορίζουμε επειδή είσαστε ε, ενθουσιώδης οπαδός των εργασιών της Επιτροπής μας, της εσωτερικής αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή. Σας δίνω λοιπόν το λόγο και κατόπιν θα ακούσουμε έναν γύρο ερωτήσεων από τους συναδέλφους μας. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, κύριε και κύριοι, προτού να μπω σε λεπτομέρειες για τα διάφορα θέματα, θα ήθελα να σας δώσω μια γενική εικόνα του τι θα ήθελα να πετύχω κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας μας στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, διότι νομίζω ότι έχουμε πολλά να μάθουμε από την οικονομική κρίση και τώρα έχει έρθει η ώρα να ε, ανταποκριθούμε. Ε, κάποια από τα μαθήματα αυτά είναι προφανή, είναι η πιο στενή συνεργασία στον τομέα της ε, οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής ε, λόγω των ανισορροπιών που υπάρχουν. Υπάρχουν όμως και λιγότερο προφανή εξίσου σημαντικά μαθήματα όμως να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε τρία βασικά σημεία. Καταρχήν, όταν επικεντρωνόμαστε στην ε, οικονομική σταθερότητα δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ε, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα. Ε, γενικά πιστεύετε ότι χωρίς αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε τις ανισορροπίες που υπάρχουν. Δεύτερον, ε, υπάρχει μια νέα σειρά πηγών για την ανάπτυξη, η καινοτομία η ε, έξυπνη αντιμετώπιση των, ε, του ανθρώπινου και φυσικού δυναμικού μας ε, και ένα πιο πράσινο μέλλον. Ε, τρίτον, ε, δεν ε, θα πρέπει να απεμπολίσουμε την αρχή ότι θα πρέπει να είναι βιώσιμη η ανάκαμψη και η ανάπτυξη. Προφανώς μπορεί να εξάγει κανείς πολλά άλλα συμπεράσματα από την κρίση. Μπορούμε όμως αυτά να τα συνοψίσουμε σε μία πρόταση. Τα οικονομικά προβλήματα ποτέ δεν ξεκινάνε από την οικονομία. Ε, γενικά ξεκινάνε από την πολιτική και την ανθρώπινη φύση. Ούτε ε, τελειώνουν με την οικονομία. Χρειάζονται λοιπόν ε, πολιτικές απαντήσεις, πολιτικές λύσεις και από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναζητώντας σωστές λύσεις, η βασική πρόκληση νομίζω ότι είναι να βλέπουμε και το δάσος και τα δέντρα ταυτόχρονα εμείς οι Ευρωπαίοι χρειάζεται να έχουμε το μεγάλο όραμα, αλλά να βλέπουμε και τις λεπτομέρειες. Ε, Κοιτώντα το δάσο, ε, λοιπόν, έχουμε ένα φιλόδοξο όραμα, την Ευρώπη 2020, που είναι κάτι παραπάνω από διάδοχο της στρατηγική τη Λισαβόνα. Είναι πιο επικεντρωμένη, είναι πιο στοχευμένη, ε, χρησιμοποιεί πιο ακριβή μέτρα, πιο ισχυρή διακυβέρνηση και κυρίως υπάρχει προοπτική μεταρρύθμιση και σε ευρωπαϊκό και επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών. Αν κοιτάξουμε τι λεπτομέρειες, τα δέντρα δηλαδή, έχουμε τον οδικό χάρτη, ο οποίος ε, θα ε, παρέχει μια πιο ισχυρή εκ των υστέρων ε, διάσταση για, την για τον οικονομικό συντονισμό. Η ΕΚΟΦΗΝ έχει ηγετικό ρόλο και άλλες ομάδες του Συμβουλίου όμως παίζουν ρόλο. Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ε, θα διεξάγει συζήτηση στρατηγική με βάση τα αποτελέσματα τη ετήσια έκθεσης ανάπτυξη ε, και τους προσανατολισμούς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ε, στόχος μας είναι να φροντίσουμε να υπάρχει συνοχή με κάποιες βασικές πρωτοβουλίες όπως είναι η Ένωση Καινοτομίας. Βλέπουμε λοιπόν τις λεπτομέρειες στα στα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο. Κάποια από αυτά συζητιούνται εδώ και πολύ καιρό, αλλά ε, πιο πρόσφατα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν από εμά να σπάσουμε το αδιέξοδο, να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο και να εισάγουμε νέες λύσεις ε, σε ε, στις πρόσφατες προκλήσεις. Κυρίες και κύριοι, όσον αφορά το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, να αναφέρω δύο βασικές αρχές, τις οποίες θα ήθελα να ακολουθήσω κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας και που πιστεύω ότι είναι σημαντικές ε, για να ε, μπορέσει να ανακάμψει η Ευρώπη. Η πρώτη βασική αρχή μου είναι η εξής οι επιχειρήσεις ε, να έχουν λιγότερες δαπάνες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αν εξαλείψουμε τα εμπόδια και δώσουμε τη δυνατότητα στις ε, επιχειρήσεις να λειτουργούν με λιγότερα έξοδα, αυτό θα βοηθήσει να ανακάμψουμε πιο γρήγορα από την κρίση, να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη. Δεν χρειαζόμαστε πιο λεπτομερή ρύθμιση, χρειάζεται να άρουμε τα εμπόδια. Οι επιχειρήσεις δημιουργούν αξία. Ε, κάποια πράγματα όμως εξεφεύγουν από αυτό το βασικό στόχο το να ε, βρίσκει κανείς το δρόμο του στους λαβυρίνθους της γραφειοκρατίας, ε, το να συμπληρώνει κανείς έντυπα, το να, η επίλυση διαφορών. Όλα αυτά είναι σπατάλη δυναμικού. Ε, αυτοί που ασκούν πολιτική λοιπόν θα πρέπει πάντα να αναρωτιόνται. Οι δράσει μα βοηθούν τι επιχειρήσει να δημιουργήσουν προστιθεμένη αξία. Υπάρχουν κάποια θέματα επιτάπητο όπου έχουμε καλές, ε, καλή δυνατότητα να απαντήσουμε με ένα σαφέ ναι. Να σα απαντήσω τρία ε, βασικά θέματα. Ε, η πράξη τη ενιαία αγορά σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή ε, πολιτική θα πρέπει να ε, αυξήσει τις ε, προσπάθειές της για να μειώσει το κόστος για τις επιχειρήσεις. Η καινοτομία θα πρέπει να γίνει λιγότερο ακριβή και να, είναι, και να διευρυνθεί η αγορά ιδεών. Επίσης, το καθεστώς της Ευρωπαϊκής εταιρεία θα εξυπηρετήσει την άρση των διασυνοριακών εμποδίων δεν ε, μπορούμε να ε, ε, εποφεληθούμε από το δυναμικό της ενιαίας αγοράς εάν οι αγορές είναι κατακαιρματισμένες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πολιτικές ώστε να αντιμετωπίσουμε τον κατακαιρματισμό των αγορών, το ετιστρέβλωση και να στηρίξουμε την κοινότητα σε όλη την Ευρώπη. ο, ήδη από τον Άνταμ Σμιθ γνωρίζουμε ότι η κατανομή της, των εργασιών ε, είναι η πηγή παραγωγικότητας ε, θέσεων εργασίας και πλούτου. Ε, ξέρουμε όμως ότι η κατανομή της εργασίας περιορίζεται από το εύρος της αγοράς. Ο κατακαιρματισμός των αγορών είναι πηγή διαφόρων αρνητικών συνεπειών είναι κάτι που εμποδίζει τις επενδύσεις και την ε, ε, δημιουργία θέσεων εργασίας. Με άλλα λόγια, ο κατακαιρματισμός της αγοράς ε, σημαίνει μείωση της δυνατότητάς μας ε, για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Με το ρυθμιστικό πλαίσιο, οι πολιτικοί θα πρέπει να αναρωτιόνται. Οι δράσεις μας αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του κατακαιρματισμού της αγοράς ή όχι. Και εδώ υπάρχουν κάποια θέματα όπου μπορούμε να απαντήσουμε με ένα σαφές ναι. Η κινητικότητα των αγαθών και υπηρεσιών ε, σε διασυνοριακό επίπεδο ε, θεωρείται μία από τις βασικές ελευθερίες στην Ευρώπη και ε, χρειάζονται και άλλες ευφυείς πολιτικές ώστε να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό της αγοράς, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες. Σωστή και συνεπής εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες σε όλα τα κράτη-μέλη αποτελεί ένα ζωτικό βήμα προς μια λειτουργική ενιαία αγορά όσον αφορά την ελευθερία παροχής υπηρεσιών σε διασυνοριακό επίπεδο. Δεύτερον, ε, η Ευρώπη σήμερα χρειάζεται ένα πλαίσιο ε, προτύπων της αγοράς που να βρίσκουν τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στο ευρωπαϊκό και εθνικό ε, επίπεδο. Επίσης θα πρέπει να, τα πρότυπα αυτά να είναι εύχριστα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μην επιφέρουν πλέον κόστος. Η αύξηση της διαφάνειας στην αγορά και η συγκρισιμότητα ε, ενισχύει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ε, να επανέλθω όμως ε, στο, στο θέμα των επιχειρήσεων με λιγότερε δαπάνε μέσα στην Ευρώπη. Ας ξεκινήσω από το Single Market Act, την πράξη τη αγοράς. αγορά. η ενιαία αγορά είναι οικονομικά η καρδιά και η ουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πλεονεκτήματα μιας μεγάλης αγοράς 500 εκατομμύρων ανθρώπων είναι οικονομικά σαφή, ωστόσο για να κεφαλοποιήσει κανείς τα πλεονεκτήματα αυτά χρειάζονται δράσεις. Δράσεις ώστε να υπάρχει ελεύθερη αγορά, ε, διευρυμένες επιλογές ε, και για να έρθουν ε, τα εμπόδια. Επιπλέον, η τεχνολογία προοδεύει με τρομερή ταχύτητα και διαμορφώνει τη ζωή μας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η ενιαία αγορά λοιπόν είναι επίκαιρο θέμα. Η 20η επέτειος της ε, ενιαίας αγοράς το 2012 προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία. Έτσι η Ουγγρική Προεδρία σκοπεύει να δώσει προτεραιότητα στην Single Market Act παρακολουθώντας ε, προσεκτικά την ε, δημόσια διαβούλευση που έχει ξεκινήσει η Κομισιόν με την ανακοίνωσή τη. και καθοδηγώντας το Συμβούλιο Υπουργών ώστε να δώσει κατευθυντήρες γραμμέ στην Κομισιόν ε, τον Μάρτιο με πληροφορίες από την Κομισιόν και πιθανότατα στον Μάιο με ε, συμπεράσματα του Συμβουλίου. Προσλέπουμε στην καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να αντιμετωπίσουμε τα σημεία συμφόρησης της ενιαίας αγοράς προωθώντας την <coughs> νομοθετική εργασία. Ε, επίσης ε, προσβλέπουμε στην υιοθέτηση των ε, τριών κοινοβουλευτικών εκθέσεων για το πακέτο της ενιαίας αγοράς. Το δεύτερο θέμα είναι το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνία. Προτείνοντα μια νέα στρατηγία για την ενιαία αγορά, ο καθηγητής Μάριο Μόντι στην έκθεσή του τονίζει ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία για ότι η μη συμφωνία για ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ε, ευρεσιτεχνία είναι ένα από τα βασικότερα κενά τη ενιαία αγορά. Ε, μετά από σχεδόν τρει ε, δεκαετίε τώρα έχουμε μια ιστορική ευκαιρία και θα πρέπει να την αδράξουμε. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι στη ζωή συχνά καθυστερούμε, αλλά ο χρόνο δεν σταματάει. Ο χρόνο που περνάει ε, ε, χάνεται. Θα ήθελα να ε, παραθέσω τη δήλωση της Άγγελα Μέρκελ ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τον πλούτο μας στην Ευρώπη, την ευημερία μας μόνο εάν είμαστε ένα, μία από τις πιο καινοτόμες περιφέρειες στον κόσμο. Συμφωνώ ότι με ένα ενιαίο σύστημα διπλωμάτων ευρωστεχνίας το οποίο θα παρέχει νομική βεβαιότητα και μειωμένο κόστος εάν δεν έχουμε ένα τέτοιο σύστημα δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε το φιλόδοξο στόχο μας τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι κάτι παραπάνω από τρόπο να κεφαλοποιήσουμε τα, τις καινοτομίες στην Ευρώπη με κάποιο, κατά κάποιο τρόπο. αντιπροσωπεύει το δικαίωμα ενός ανθρώπου ε, στα προϊόντα ε, του νου του. Γι' αυτό η Ουγγρική Προεδρία θα επιδιώξει να πετύχει το στόχο αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα. Καθότι η τελική απόφαση για ε, το ενιαίο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνία πρέπει να λυθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα και ε, εάν η διευρυμένη συνεργασία είναι η μόνη λύση για να επιτευχθεί αυτό, εμεί ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε τη διαδικασία αυτή. Ταυτόχρονα ζητούμε ευγενικά από το Κοινοβούλιο να συνενέσει ώστε να δώσει τη δυνατότητα στο Συμβούλιο να εγκρίνει τη διευρυμένη συνεργασία στο Συμβούλιο ανταγωνισμού στις αρχές ε, Μαρτίου. Θα μπορέσουμε τότε να ξεκινήσουμε τη δουλειά μας με βάση την πρόταση της Κομισιόν ε, πάνω στις ρυθμίσεις, ε, τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του ενιαίου διπλώματο τεχνίας και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια στη συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά τις, ε, την μετάφραση, στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα γλωσσικό καθεστώς το οποίο να βασίζεται στις τελευταίες ε, προτάσεις της Κομισιόν. Επίσης έχουμε το θέμα της Ευρωπαϊκής ε, Εταιρείας, Μεταρχικής Εταιρείας. Αυτό το θέμα έχει μακρά ιστορία. Αυτή η νέα νομική οντότητα θα επιτρέψει στους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν εταιρείε τη ίδια μορφή, άσχετα από το αν ε, δραστηριοποιούνται στο δικό του κράτο μέλο ή σε άλλο. Ε, ακολουθούμε την ε, σουηδική πρόταση του Δεκεμβρίου 2009 ε, που πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει βάση για συμβιβασμό και στόχος μας είναι, στο βαθμό που είναι δυνατόν, να μην ξανανοίξουμε τη συζήτηση παρά μόνο για τρία βασικά θέματα. Το θέμα της έδρας, ε, των ελάχιστων κεφαλαιοκάνω απαιτήσεων και την ε, συμμετοχή των εργαζομένων. Η Ουγγρική Προεδρία θα ήθελε να καταβάλει προσπάθειες ώστε να πετύχουμε συμβασμό στα θέματα αυτά. Και κύριοι, περνάω στην επόμενη, στη δεύτερη αρχή μου, ε, την αντιμετώπιση του κατακαιρματισμού της αγοράς. Ε, να σας ε, δώσω μερικά στοιχεία για το πιο σημαντικό φάκελο στον οποίο μπορούμε να προωθήσουμε τα πράγματα. Έχουμε την, υπηρεσία, την οδηγία της υπηρεσίας. Μία από τις πιο κατακαιρματισμένες αγορές είναι αυτή των υπηρεσιών, ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με τη νέα τεχνολογία. Παρότι ο τομέας των υπηρεσιών αντιπροσωπεύει το 70% του ΑΕΠ στην Ευρώπη, η αγορά υπηρεσιών είναι πολύ κατακαιρματισμένη και σύμφωνα με, το, με την έκθεση Μόντι, μόνο το 20% των υπηρεσιών που παρέχονται έχουν διασυνορική διάσταση. Έτσι υπάρχει ένα ε, κενό παραγωγικότητας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει διευρυνθεί την τελευταία δεκαετία. Και υπάρχει ε, ε, ζημιά στην οικονομική ανάπτυξη, καθότι σύμφωνα με, την, με τους υπολογισμούς για την εφαρμογή της Οδηγίες για τις υπηρεσίες ε, υπάρχει... η, εφαρμογή αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση 0,6 με 1,5% του ΑΕΠ. Όσον αφορά την ε, οδηγία για τις υπηρεσίες, ε, καταλαβαίνω ότι θα ψηφίσει η ΜΚΟ την σχετική επιτροπή για την εφαρμογή της αμέσως μετά από την ομιλία μου. Θα συνεργαστούμε στενά με την Κομισιόν για να παρακολουθήσουμε τα αποτελέσματα της ε, αμοιβαία αξιολόγησης ε, όσον αφορά την ε, εφαρμογή της οδηγίας. Στόχος μας είναι να προτείνουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου με βάση την ανακοίνωση της Κομισιόν, ώστε η εφαρμογή της οδηγίας αυτής να παραμείνει ψηλά στην ατζέντα των κρατών μελών ε, σε θέματα ε, ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Επίσης, όσον αφορά την τυποποίηση, ανάλογα με την ε, ημερομηνία διαβίβασης της ανακοίνωσης και της νομοθετικής πρότασης της Κομισιόν, η Ουγγρική Προεδρία θα ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ομάδας εργασίας ε, για το θέμα της τυποποίησης. Η Προεδρία επίσης ε, θα βρίσκεται σε επαφή με τους συνομοθέτες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ε, συνεργαστεί στενά με τις επόμενες Προεδρίες. Η πρόταση αναμένεται το, την άνοιξη του 2011 και θα συνοδεύεται από ανακοίνωση της Κομισιόν πάνω στο ίδιο θέμα θα τροποποιεί το πλαίσιο πολιτικής τυποποίησης όσον αφορά την νομική πλευρά, θα δώσει όμως και πολιτικά μηνύματα όσον αφορά την ε, σημασία της ε, αποτελεσματικής ετυποποίησης ως, ε, ως μέσο για την εναρμόνιση και την διευκόλυνση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων στην Ευρώπη. Τα πρότυπα επίσης θα πρέπει να πληρούν κάποια κοινωνικά κριτήρια ή περιβαλλοντικά κριτήρια. Επίσης έχουμε την οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Ο Χέρπερτ Χούβερ, πρόεδρος, ε, κατά την, ε, πρόεδρος της Αμερικής κατά τη διάρκεια της ε, μεγάλης κρίσης, έλεγε, είπε κάποτε ότι η ότι ο ανταγωνισμός ε, δεν, είναι μόνο, δεν προστατεύει μόνο τον ε, καταναλωτή, αλλά αποτελεί και κίνητρο για την πρόοδο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να ε, επιδείξουμε τη διαφορά ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι πεπισμένο ότι όλοι οι στόχοι για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και διατήρηση του υψηλού επίπεδου προστασίας των καταναλωτών χωρίς να ε, επιβάλλουμε ε, περιττό διοικητικό άχθος ε, στις εταιρείες. Αυτά μπορούμε να τα πετύχουμε ταυτόχρονα και αυτό αποτελεί ένα από τα βασικότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό η Ουγγρική Προεδρία πιστεύει ότι μετά από σχεδόν δυόμιση χρόνια διαπραγματεύσεων έχει έρθει η ώρα να πετύχουμε συμφωνία πάνω στην οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Ιδιαίτερα φιλοδοξία της Προεδρίας είναι να πετύχουμε συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Προεδρία θα παρακολουθεί στενά τις συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην ΙΜΚΟ και την Επιτροπή Τζούρι και θα βρίσκεται σε επαφή με τον εισηγητή κύριο Σφάπ για να συμφωνηθεί ε, ένα ε, χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις κατά την πρώτη ανάγνωση. Όσον αφορά το επίπεδο εναρμόνισης, η Προεδρία στοχεύει στην εξέβρεση ε, πρακτικών λύσεων που να βασίζονται ε, στον συνδυασμό ελάχιστης και μέγιστη εναρμόνιση, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, όσον αφορά του στόχου της ε, οδηγίας. Κυρίες και κύριοι, Σήμερα η Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις που απαιτούν σημαντικές προσπάθειες από όλους μας. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πιο ταπεινή φιλοδοξία από την ενίσχυση της, Ευρωπαϊκής, ενίσχυση της Ευρώπης. Αυτό είναι ε, το σύνθημα της Ουγγρικής Προεδρίας. Η ευρωπαϊκή κοινότητα ανήκει σε όλα τα μέλη της ε, και θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τα, τις παραδόσεις και τις ε, φιλοδοξίες όλων των μελών της. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Μάργαρετ Θάτσερ σε μια από τις πιο σημαντικές ομιλίες στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για την ομιλία της στην το 1988. Παρότι θα πρέπει να διευρύνουμε τον ορίζοντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκει σε όλους τους πολίτες της και θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις παραδόσεις και τις φιλοδοξίες, τις ελπίδες όλων των πολιτών της επίσης. Πιστεύω λοιπόν ότι το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεργάζονται στενά. Εάν ε, συνεργαστούμε, θα έχουμε τι ε, καλύτερε δυνατότητε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Αν μπορέσουμε να πετύχουμε κάποια βασικά βήματα ώστε να μειώσουμε το κόστο για τι επιχειρήσει και να εμποδίσουμε τον κατακαιρματισμό των αγορών, θα συμβάλλουμε στην ανάκαμψη τη Ευρώπη. Κυρίε και κύριοι, να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου στους, ε, στην Ισπανική και Βελγική Προεδρία και προηγούμενες προεδρίες για την εξαιρετική δουλειά που κάνανε σε συνεργασία μαζί σας στον, τομέα της ε, πολιτικής ανταγωνισμού όσον αφορά για παράδειγμα την ελεύθερη κινητικότητα αγαθών υπηρεσιών και ε, στον τομέα των ε, δικαιωμάτων των καταναλωτών. Να τονίσω την αφοσίωση της Ουγγρικής Προεδρίας να συνεχίσει την δουλειά της στο πνεύμα αυτό. Ε, και εσεί είσαστε βασικό παράγοντα ε, στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Ε, οι αρμοδιότητες σα ενισχύθηκαν με την συνθήκη της Ε, Θα συνεργαστούμε και στα πλαίσια του τρίου με του Πολωνούς και Δανού συναδέλφους μα για να συμπληρώσουμε τη δουλειά των Ισπανών και Βέλγων συναδέλφων. Αυτή ήταν η εισαγωγή μου με λίγα λόγια. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ε, πολύ ευχαρίστω θα απαντήσω στις ερωτήσεις και παρατηρήσεις σας. Uh, Κύριε Υφυπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε για τις ξεκάθαρες εξηγήσεις που δώσατε για τις προτεραιότητές σας. Και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι ότι θα γίστε ο ίδιος της ε, αρμόδιας επιτροπής του Συμβουλίου και ότι θα αναλάβετε ευθύνη για τις προτεραιότητες στις οποίες αναφερθήκατε. Γνωρίζετε πολύ καλά λοιπόν ποιες είναι οι βασικές εργασίες της δικής μας κοινοβουλευτικής επιτροπής και Βλέπετε ότι μαζί μας ε, έχουμε τον εισηγητή για την ε, τυποποίηση, ο οποίος έκανε την ε, έκθεση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η κυρία Γκέπχαρτ είναι η αρμόδια για την οδηγία για τις υπηρεσίες, έκθεση την οποία θα ψηφίσουμε σήμερα σύντομα. Ελπίζω λοιπόν ότι θα έχετε την ε, δυνατότητα να προσκαλέσετε κάποιους από τους ηγητές μας να συναντήσουν και κάποιους από τους συναδέλφους σας στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας προκειμένου να καταφέρετε να τους μεταδώσετε προς όλους την δυναμικότητα αυτή που εμείς έχουμε εδώ πέρα όσον αφορά τις προτεραιότητες στις οποίες αναφερθήκατε. Θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε τώρα ερωτήσεις ε, σε ομάδες των τριών. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να απαντήσετε κιόλα. Να είστε σύντομοι σας παρακαλώ πολύ. Θα ζητήσω από τα μέλη από την κάθε μία από τις πολιτικές ομάδες που είναι εδώ να πάρουν το λόγο Σβάμπ, Γκέπχαρτ και Κρότσμαν η πρώτοι. Κύριε Σβάμπ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Τσεβάλφε, χαίρομαι πολύ που τόσο νωρίς στην Ουγγρική Προεδρία καταφέρατε να έρθετε και να μας μιλήσετε εδώ πέρα και Χαίρομαι πολύ που έχετε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά για τα ζητήματα τα οποία μας αναφέρετε. Σας ευχαριστώ επίσης που είπατε ότι θα συνεργαστείτε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι καθοριστικό όσον αφορά τα ουσιώδη ζητήματα που εμεί έχουμε στις προτεραιότητές μας. Εμείς, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλαμε τα θέματα αυτά να βρίσκονται πραγματικά στην πρώτη γραμμή. Αναφερθήκατε στην δράση την οποία θα αναλάβετε και έχουν ληφθεί κάποιες σημαντικές αποφάσεις και τοποθετήσεις όσον αφορά συγκεκριμένα ζητήματα όπως το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Βρεσιτεχνίας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια συζητάμε το ζήτημα αυτό και επιτέλους τα πράγματα κινούνται. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ελπίζουμε πραγματικά ότι θα καταφέρετε να προωθήσετε το θέμα αυτό. Μιλήσετε επίσης για τον κατακαιρματισμό στην εσωτερική αγορά και αυτό το ζήτημα μας έχει απασχολήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρέπει επιτέλους να ληφθεί δράση και στηριζόμαστε σε εσά. Τρίτον, πράξη ενίας αγοράς ένα σημαντικότατο πλέον τμήμα της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Αναφερθήκατε στην ευημερία, αναφερθήκατε στη δήλωση της κυρίας Μέρκελ. Θεωρώ τα στοιχεία αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά προκειμένου να σημειώσουμε πρόοδο. Αναφερθήκατε επίση στην οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είμαστε ευγνώμονε που το Συμβούλιο έχει εργαστεί για το ζήτημα αυτό πολύ σκληρά και ότι καταφέρατε τελικά να σημειώσετε πρόοδο. Εμεί σύντομα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσουμε για το ζήτημα αυτό και μετά την ψηφοφορία θα είμαστε θέση να γνωρίζουμε πόσο χρόνο θα χρειαστούμε προκειμένου να καταλήξουμε στην οριστική τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορώ να σα πω όμω αυτή τη στιγμή ότι Ελπίζουμε να εγκρίνουμε το νομοθέτημα αυτό για τα δικαιώματα των καταναλωτών το σημαντικότερο δυνατό και ελπίζουμε γρήγορα να επιθυμεί να κινηθεί και το Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή ψηφίσει το Κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω ότι θα καταφέρει το Συμβούλιο γρήγορα να ακολουθήσει και αυτό με μια δική του έγκριση. Η κυρία Γκέπχαρτ, σα ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την ε, πολύ καλή αυτή παρουσίαση που κάνατε όσον αφορά τις ε, προθέσεις σας ε, στα πλαίσια της ε, Ουγγρικής ε, Προεδρίας. Συμφωνούμε σε πάρα πολλά σημεία. Η ε, δική μου πολιτική ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών βασίζεται σε εσά προκειμένου να καταφέρουμε μέσω μια επικοδομητική συνεργασία να ξεπεράσουμε τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο εμπόριο και γενικότερα στην εσωτερική αγορά. Ελπίζω θα καταφέρουμε λοιπόν να συνεργαστούμε επικοδομητικά για να πετύχουμε όλα αυτά τα οποία, στα οποία αναφερθήκατε. Θεωρώ ότι η προσέγγιση σα είναι πολύ καλή Θεωρώ και εγώ ότι θα πρέπει να περιοριστούμε περισσότερο σε πράξεις και να μην αναλωθούμε πάρα πολύ σε λόγια και θεωρητικές προσεγγίσεις. Είμαι η συγγήτρια για την οδηγία της υπηρεσίας στην οποία αναφερθήκατε. Το να ληφθεί δράση για το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχουμε συνομιλητές συνεργάσιμους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε επίση τι έχει γίνει στα κράτη-μέλη. Κάθε φορά που μιλάμε για το γεγονός της αμοιβαία αναγνώρισης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι συντονισμό υπάρχει ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Μέσω αυτού του μέσου θα καταφέρουμε ουσιαστικά να εξασφαλίσουμε ότι οι εταιρείε, οι επιχειρήσει και οι καταναλωτέ θα έχουν την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στην αγορά. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και η δική μου πολιτική ομάδα βρίσκει πολύ καλό το ότι θέλετε να ασχοληθείτε με το θέμα του Ευρωπαϊκού ε, Διπλώματο Ευρεσιτεχνία, διότι αυτό είναι κάτι απαραίτητο μέσα στην Ευρώπη. Έτσι μπορούν να εξοικονομηθούν πολλά χρήματα για την καινοτομία. Ε, έχω όμως ένα αλλά, κύριε Πρόεδρε. Ε, στον ε, τομέα των δικαιωμάτων των καταναλωτών συμφωνώ μαζί σας. Θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, αλλά η ποιότητα έχει πιο μεγάλη σημασία από την ταχύτητα. Σημασία μεγάλη, λοιπόν, έχει η διαφάνεια. Και στο θέμα αυτό... Σημαντικό είναι να ασχοληθούμε με βασικά θέματα όπως το, το τα δικαιώματα των καταναλωτών και να μην το κάνουμε αυτό βιαστικά. Η δική μου πολιτική ε, ομάδα δεν θα συμφωνήσει με κανέναν τρόπο σε συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση. Σας το λέω αυτό ήδη σήμερα για να μην ε, τρέφετε αυταπάτες. Ε, θέλουμε διαφάνεια. Η πολίτες, ε, οι καταναλωτές έχουν ε, δικαίωμα να γνωρίζουν τη διαπραγματευτική βάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέναντι στο Συμβούλιο των Υπουργών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και γι' αυτό πρέπει να σας ε, πω ότι έτσι έχουν τα πράγματα και ελπίζω κύριε εισηγητή να μην έχετε στόχο να ε, κάνετε διαπραγματεύσεις ήδη τώρα. Ε, αυτό δεν θα ήταν τίμιο. Δεν περιμένω όμως να κάνετε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ακούσαμε αρκετά θέματα ε, στα οποία έχει να απαντήσει ο Υπουργός. ο κύριος Κρότσμαν. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ μιλήσατε για πράγματα που ενδιαφέρουν πολύ ε, την ομάδα των φιλελευθέρων. Είπατε τι πρέπει να γίνει για να ε, υπερνικήσουμε την κρίση. Είπατε ότι πρέπει να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι ε, ε, παράγουμε προϊόντα όχι μόνο για την ε, ευρωπαϊκή αγορά αλλά και για την παγκόσμια αγορά. Τα ε, προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη θα μπορούσαμε να τα εξάγουμε μόνο αν οι τιμές είναι ανταγωνιστικές. Αναφερθήκατε και στην καινοτομία. Σε σχεδόν όλα τα κράτη της Ευρώπης, αλλά ιδιαίτερα στη Γερμανία, έχουμε πολύ ψηλό κόστος σε κάποια θέματα. Μόνο λοιπόν με καινοτόμα προϊόντα θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε στην ε, παγκόσμια αγορά και όχι με φτηνά προϊόντα. Και τα άλλα κράτη-μέλη θέλουμε να τα ενθαρρύνουμε να ε, ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Στην ε, Γερμανία συζητάμε τη, τη συμβολή της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ. Ε, και το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν το 1 τρίτο. Ε, αν ε, τα άλλα κράτη-μέλη επιδιώκουν μια συμβολή κατά 10% της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ. Βλέπουμε ότι θα πρέπει κάποια κράτη-μέλη να κάνουν κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικά. Ε, η ανταγωνιστικότητα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ε, ο το στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας ε, για τον κόσμο. Παράκλησή μου αναφερθήκατε στην Single Market Act και θα ήθελα να συνδέσω το, το θέμα αυτό με την κριτική μας στάση βλέπουμε όλο και περισσότερα σε κάποια κράτη-μέλη ε, ο κόσμος να είναι επιφυλακτικός απέναντι στην Ευρώπη. Ε, ακριβώς αντίστροφα είναι τα πράγματα, όμως ε, η Ευρώπη μας έχει δώσει ένα μακρό διάστημα ειρήνης και αυτό από μόνο του σημαίνει ότι η Ευρώπη αξίζει τον κόπο, αλλά έχει ωφελήσει πολύ τα κράτη και οικονομικά. Η Ευρώπη είναι ε, από τις πρώτες χώρες στις εξαγωγές αλλά και στις εισαγωγές. Στην ε, βιομηχανία μας λοιπόν ε, πολύ συχνά παράγουμε κάποια ημιτελή ή με κατέργαστα προϊόντα. Είπατε ότι θέλετε να μειώσετε το κόστος για τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να φροντίσουμε οι παραγωγή να είναι λιγότερο ακριβή. Μία ερώτηση. Η Ουγγαρία έχει αυξήσει τους φόρους που είναι επίσης κόστος για τις επιχειρήσεις. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, θα σας δώσω την ευκαιρία να απαντήσετε σε αυτές τις τρεις παρεμβάσεις. Έχω έξι ομιλητές. Ε, θα έχουμε λοιπόν άλλους δύο γύρους των τριών ομιλητών. Υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Ωραία. Στον επόμενο γύρο ο κύριος ε, Κόσνη και ο κύριος Τριανταφυλλίδης και ο κύριος Καμιέσκη. Ο κύριος ε, Ντεκάμπος, η κυρία Κορατσαμπίλ και η κυρία Στάιλερ. Ε, κύριε Υπουργέ, μπορείτε να απαντήσετε. Uh, uh, uh, Μάλλον θα μιλήσω την μητρική μου τη γλώσσα για να απαντήσω σε ερωτήσεις αυτές. Στα γερμανικά συμφωνώ απόλυτα κύριε Σβάπ με αυτά που λέτε. Χρειαζόμαστε δράσεις, ε, χρειαζόμαστε ε, συγκεκριμένα πράγματα για να μπορέσουμε να προωθήσουμε, την, ε, να τις διαδικασίες. Στην αρχή όταν είδα τους φακέλους αυτούς είδα όχι μόνο τον μεγάλο αριθμό των θεμάτων που υπάρχουν, είδα ότι σε πολλές περιπτώσεις μιλάμε για ιστορικό πολλών ετών και το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Ε, ακριβώς σε αυτήν την ε, περίοδο της ε, κρίσης δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε περισσότερο τους φακέλους αυτούς που έχουν πίσω τους ιστορία 5-10 ετών. Χρειαζόμαστε λοιπόν και τη στήριξη του Κοινοβουλίου. Όσον αφορά τη μείωση των ρυθμίσεων, που, αναφέρει, που ανέφερε η κυρία Κέπχαρτ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Όταν βλέπουμε πού βρισκόμαστε ε, σήμερα, ε, θέλουμε να κινητοποιήσουμε τις επιχειρήσεις. Ε, ωστόσο ζούμε σε εποχή ε, εξοικονομήσεων. Ε, Πώ μπορούμε να βοηθήσουμε χωρίς χρήματα, με λιγότερη ρύθμιση. Θέλουμε λοιπόν να απαλλάξουμε τις επιχειρήσεις από ένα μεγάλο βάρος και γι' αυτό είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε το θέμα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και γι' αυτό βιαζόμαστε λίγο όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα και στην ταχύτητα. Ε, αλλά Λόγω της κατάστασης που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ήδη η πρώτη ανάγνωση θα αποτελούσε μια καλή λύση και έτσι θα προωθήσουμε το έργο. Ελπίζω να μην ε, γίνει αυτό εις βάρος της ποιότητας. Ε, θα φροντίσουμε να παραμείνει υψηλή η ποιότητα, αλλά βρισκόμαστε υποχρονική πίεση. Η Ευρώπη περιμένει από μας ε, πράξεις έργα και θέλουμε να προωθήσουμε, θέλουμε να πετύχουμε πρόοδο σε θέματα που έχουν πίσω τους ιστορία πενταετίας ή δεκαετίας όσον αφορά τη βιομηχανία και την παροχή υπηρεσιών. Σε κάποιες χώρες ε, οι υπηρεσίες έχουν περισσότερο βάρος, σε άλλες ε, η βιομηχανική παραγωγή. Στην ε, κρίση είδαμε ότι οι χώρες και οι περιφέρειες που είχαν ισχυρή βιομηχανική βάση επιβίωσαν καλύτερα στην κρίση. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και στην εποχή της ε, παγκοσμιοποίησης της, ε, της ε, κοινωνίας των υπηρεσιών το να παράγει κανείς κάτι αυτό είναι σημαντικό. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το έχουμε κατά νου. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε την παραγωγή αυτή. τέθηκε μια ερώτηση για την Ουγγαρία. και θα ήθελα να πω σε αυτό το θέμα ότι κάνουμε και τα δύο. Δηλαδή η ουγγρική πολιτική ε, δεν ε, είναι mainstream εδώ. Με το ένα χέρι μειώνουμε τη φορολογία, με το άλλο αυξάνουμε κάποιους φόρους. Μετά από την μεταπολίτευση ε, κληρονομήσαμε μία μαύρη τρύπα στα στην ε, ε, κρατική οικονομία και για να ε, μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό έπρεπε να επιβάλλουμε έναν φόρο της κρίσης. Μειώσαμε τον εταιρικό φόρο από 19% σε 10% φέτος θα εισπράξουμε έναν ενιαίο φόρο flat tax και ελπίζουμε έτσι να μπορέσουμε να ε, δώσουμε ορμή στην ε, οικονομική ζωή και ο φόρος κρίσης αυτός έχει χρονικό περιορισμό τρία χρόνια, πέρσι, ε, φέτος και του χρόνου. Ελπίζουμε ότι τα άλλα πράγματα που έχουμε κάνει για να δώσουμε ορμή στην οικονομία, η μείωση των φόρων και η μείωση της γραφειοκρατίας και οι εξοικονομήσεις στις δημόσιες δαπάνες, ε, πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσουν να έχουμε πιο ισχυρή οικονομική ανάπτυξη από ό,τι κατά τα άλλα. Και έτσι μετά το 2012 δεν θα χρειαζόμαστε πια αυτόν τον ε, φόρο κρίσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Τώρα αν μπορούμε να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε ακόμα ένα τέταρτο περίπου. Θέλω να ενθαρρύνω του συναδέλφου να είναι συνοπτικοί. Ο κύριε Κόσμη, κύριε Τριανταφυλλίδης, στη συνέχεια κύριε Κόσμη, καταρχήν. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, θα είμαι πολύ σύντομος εκπροσωπούμε διαφορετικέ πολιτικέ ομάδε. Επομένω έχουμε διαφορετικέ ε, πολιτικέ απόψει, αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε στο εξή. Και η κυρία Γκέπχαρτ και ο κύριος Γκρότσπερκ ε, και ο κύριος Βάρπ ε, το ανέφεραν αυτό. Λιγότερη γραφειοκρατία. Αν θέλουμε να έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία, λογικά θα πρέπει να έχουμε λιγότερη ρύθμιση και όχι περισσότερη. Γιατί η λιγότερη ρύθμιση προωθεί την ανταγωνιστικότητα της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η Ουγγρική Προεδρία έχει ακολουθήσει μια ενεργητική προσέγγιση απέναντι στην ευρωπαϊκή τυποποίηση, γιατί αυτό είναι υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Έτσι λοιπόν ακολουθείται μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και όχι το αντίθετο. Η δική μας Επιτροπή είναι έτοιμη να ασχοληθεί με το θέμα της τυποποίησης. Είμαστε ιδιαίτερα ενεργητικοί σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ε, γενικότερα για το θέμα της οδηγίας ε, για τα δικαιώματα των καταναλωτών να πω ότι συμφωνώ με αυτά που έχει πει η κυρία Κέμπαρτ ότι εμείς θα προτιμούσαμε να πάμε στη δεύτερη ανάγνωση για να έχουμε πλήρη διαφάνεια ε, και να ξέρουμε και τις θέσεις του Συμβουλίου. Θα προχωρήσω με δύο μικρές ερωτήσεις. Πρώτα στο θέμα της καινοτομίας. Ε, γίνεται αντιληπτό ότι στο κομμάτι της χρηματοδότησης της ε, καινοτομίας υστερούμε πάρα πολύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν δυσκολίες στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και γι' αυτό η Προεδρία λαμβάνει υπόψη αυτό το δεδομένο για να το για το σχεδιασμό του 8ου προγράμματος και ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό το σημείο ποιες δράσεις προτίθεται να αναλάβει η Προεδρία και ποιες προτάσεις έχει να καταθέσει στο τραπέζι των συνομιλιών. Και η δεύτερη μου ερώτηση έχει να κάνει με τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, για τις οποίες δεν έχω ακούσει αρκετά. Όπως λέχθηκε και στη συζήτηση της Επιτροπής, η Κομισιόν μελετά διάφορες προτάσεις για να τις καταθέσει προς συζήτηση μέσα από την Πράσινη Βίβλο. Ποιε είναι οι απόψεις και οι στόχοι της Προεδρίας σας για αυτές. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κανιέτη. Κύριε Υπουργέ, Θέλω να καλωσορίσω όλα όσα είπατε σχετικά με την επανέρεξη της πράξης της Ενίας αγοράς και της Ενίας αγοράς. Είμαι μία από τους εισηγητές ε, που συντάκτουν την έκθεση για τη διακυβέρνηση της Ενίας αγοράς. Και αν εξετάσουμε τα προβλήματα, ένα από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξα είναι ότι αν δεν υπάρχει ισχυρή υποστήριξη από τα κράτη-μέλη, ε, δεν είναι δυνατό να επαναλειτουργήσει αποτελεσματικά η νέα αγορά. Εγώ εκτιμώ την αποφασιστικότητα σας να συνεδριάσει το Συμβούλιο και να προεδρεύσετε το Συμβουλίο γύρω από αυτή τη συζήτηση. Όμως θέλω να σας ζητήσω όχι μόνο να παρακολουθήσετε στενά την δημόσια συζήτηση για την έννοια αγορά, αλλά να αφιερώσετε ιδιαίτερη ενέργεια στο να πείσετε τους συναδέλφους σας στα κράτη-μέλη να δείξουν μεγαλύτερη υποστήριξη στην ενιαία αγορά γιατί αποτελεί ατμομηχανή ανάπτυξης για την Ευρώπη. Αυτή η πράξη έχει την ίδια αξία με τη στρατηγική για την Ευρώπη για το 2020. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, να σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε σε αυτά τα τρία σημεία που αναφέραν συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ για την τυποποίηση. Ναι, η τυποποίηση είναι ένα ζήτημα και θα χαρώ πάρα πολύ αν μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Γιατί εμείς ε, χρειαζόμαστε πρώτη νομικά ασφαλή και τα πρότυπα αποτελούν ε, ένα τμήμα της μάχης για την καταπολέμηση αυτής της κατακαιρματισμένης αγοράς που έχουμε σε ορισμένα σημεία της Ευρώπης. Για να επανέλθω τώρα στο θέμα των δικαιωμάτων ε, των καταναλωτών και της πρώτης και δεύτερης ανάγνωσης. Θα προσπαθήσουμε να το επιλύσουμε αυτό το θέμα στην πρώτη ανάγνωση. Και όπως σας είπα, Κατανοώ πλήρως ότι πρέπει να το προωθήσουμε γρήγορα το ζήτημα γιατί έχει να κάνει με την ποιότητα. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία για την καινοτομία. Έχω την τιμή και την τύχη να προεδρεύω τη Επιτροπής που ασχολείται ε, με την έρευνα, την πολιτική του διαστήματος, στην ενιαία αγορά, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο να ασχοληθούμε με την πολιτική καινοτομία και τη χρηματοδότηση, αλλά θα έχουμε την ενδιάμεση έκθεση του προγράμματος ε, πλαισίου του 7ου προγράμματο πλαισίου το Μάρτιο και από εκεί θα εξάγουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα για το πώ θα χρηματοδοτήσουμε και την καινοτομία. Και επίση ε, θέλω να αναφερθώ στο ότι το κύριο ζήτημα είναι ε, πόσο ευρύ είναι η επιχειρηματική τομή και πώ καλύπτονται από την καινοτομία. Θα έχουμε και ε, μία συνάντηση σε μία πόλη κοντά στη Βουδαπέστη και θέλουμε να αφιερώσουμε μισή μέρα για να συζητήσουμε το πώ θα χρηματοδοτήσουμε την καινοτομία με έναν καινοτόμο τρόπο. Θα καλέσουμε εμπειρογνώμονε και υπουργού για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Τώρα, η πολιτική στήριξη ε, για το Single Market Act, για την πραξενή αγορά, να είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πολλές φορές ε, έχουμε εξηγήσει πόσο σημαντικό είναι να έχουμε την ενιαία αγορά. Γιατί αποτελεί την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οικονομίας. Και πάντοτε εξηγούμε τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς. Σίγουρα η πράξη της ενιαίας αγοράς περιλαμβάνει τώρα 50 διαφορετικά μέτρα και ένα από ε, τα κύρια καθήκοντα μετά από τη διαβούλευση και αφού ακούσουμε και τις δικές σας προτάσεις θα είναι να βρούμε αυτά τα 15-20 θέματα όπου θα πούμε «Α, ωραία, εδώ πρέπει να κινηθούμε το συντομότερο δυνατόν». Πρέπει να τα προωθήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και ελπίζω ότι στην ε, συνάντηση που θα έχουμε θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε αυτά τα 15 μέτρα Αυτά τα 15 μέτρα είναι ζωτική σημασίας ε, γιατί αντικατοπτρίζουν τις νέες εξελίξεις, τις νέες τεχνολογίες. Γιατί η ενιαία αγορά και ο κανονισμός ε, και η ρύθμιση, με συγχωρείτε, είναι ε, ένα συνεχιζόμενο θέμα. Οι τεχνολογίες αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή δεν μας περιμένουν εμάς. Η τεχνολογία τρέχει με το δικό της ρυθμό και έχει αλλάξει τη ζωή μας εντελώς τις τελευταίες δεκαετίες. και τι συνέβη την τελευταία δεκαετία με τις νέες τεχνολογίες. Έτσι λοιπόν ε, θα επιλέξουμε εμείς αυτά τα 15-20 θέματα, αυτούς του 15-20 φακέλους, όπου είναι σημαντικό να κινηθούμε και να σημειώσουμε πρόοδο. Νομίζω ότι ε, θα είναι πολύ σημαντικό να αντικατοπτρίζουμε στα θέματα αυτά και τις νέες τεχνολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Οι τελευταίοι τρεις ομιλητές μας, Κάμπος, Κοράτσα Μπίλτε και Στάιλερ. Κοράτσα Κάμπος πρώτα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα αγγλικά για να προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα. Σας ευχαριστώ, Υπουργέ, για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ για την πλήρη παρουσίαση που κάνατε. Θα μπορούσα να σας θέσω πολλές ερωτήσεις, τις συνοψίζω όμως σε ένα μόνο σημείο. Θα θυμάστε ότι πριν από ένα μήνα η Ιρλανδία άρχισε να ζητά οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το φορολογικό τάμπινγκ καθώς επίσης και για τον πολύ χαμηλό φόρο που υπήρχε στην Ιρλανδία για τις εταιρείες, επιχειρήσεις στην δική σας την χώρα έχετε μειώσει στο 10% τον φόρο επί των εταιριών. Αν κάθε χώρα η οποία βρίσκεται σε δινή οικονομική θέση κάνει κάτι τέτοιο, πώς θα προχωρήσουμε μπροστά, τι μπορούμε να περιμένουμε, πώς θα καταφέρουμε να πετύχουμε την απαραίτητη αλληλεγγύη από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, αν Κάθε φορά βλέπουμε ότι τελικά δεν υπάρχει φορολογική εναρμόνιση. Πρόεδρο, Σα ευχαριστούμε πολύ. Ήσασταν σύντομο και πολύ συγκεκριμένο. Κυρία Κοράτσα Μπίλτε, σα ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για την αποφασιστικότητά σας να βάλετε την πραγματική οικονομία στο κέντρο των προτεραιότητών σας. Είπατε ότι θέλετε να εξαλείψετε όλα τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και ως εισηγήτρια για την έκθεση του λιανικού εμπορίου, ενός δίκαιου λιάνου εμπορικού τομέα, θα ήθελα να σας αναφέρω τις ανησυχίες οι οποίες έχω για τα εφιστάμενα εμπόδια που υπάρχουν για την ελεύθερη κυκλοφορία και εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε να εφίστανται ακόμα τα εμπόδια αυτά. Χαίρομαι πάρα πολύ που αναφερθήκατε στην οδηγία για τις υπηρεσίες και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Προεδρία να αναλάβει δράση και να ασκήσει πίεση στα κράτη-μέλη προκειμένου να εφαρμόσουν πλήρω την υφιστάμενη νομοθεσία, ιδίω όσον αφορά την οδηγία για τι υπηρεσίε και τη δέσμη μέτρων για τα προϊόντα, για τα αγαθά. Επίση, αναφερθήκατε στη δική σας τη χώρα στο ζήτημα της φορολογίας. Σαφώς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει η αρχή της επικουρικότητας και ότι η φορολογική πολιτική είναι τελικά εθνική αρμοδιότητα. Πρέπει όμως μαζί σας και με τους συναδέλφους σας να έχουμε ένα επικοδομητικό διάλογο και να δούμε πώς οι φόροι αυτοί ενδεχομένως να επηρεάζουν τους ε, παράγοντες που έρχονται από τρίτες χώρες και πως πολλές φορές αυτή η εθνική φορολογική πολιτική δημιουργεί ένα ανισότιμο πεδίο ανταγωνιστικότητας. Επίσης υπάρχουν κάποιες άλλες νομοθεσίες σχετικά με το εμπόριο που εγκρίθηκαν πρόσφατα που και πάλι δημιουργούν τη δυνατότητα για συγκεκριμένες συμβάσεις εμπορικές που και πάλι εμποδίζουν από κάποιους οικονομικούς φορείς να συμμετέχουν ισότιμα στην εσωτερική αγορά καθότι πρέπει να προσαρμόσουν κάθε φορά το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Εμείς θα θέλαμε να μιλήσουμε με σας ανοιχτά για τα ζητήματα αυτά και ελπίζω ότι και εσείς θα θελήσετε να ανοίξετε ένα διάλογο μαζί μας. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε κυρία κράτσαμπιλτη κυρία Στάιλερ, έχει το λόγο τελευταία μιλήτρια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τι πρόκειται να κάνει η Ουγγρική Προεδρία προκειμένου να ασχοληθεί με την ψηφιακή ατζέντα και ιδιαίτερα για να κλείσει το ψηφιακό χάσμα, να αυξηθεί η πρόσβαση στην, στα ευρυζωνικά δίκτυα και πώς μπορούμε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε την απαραίτητη ψηφιακή υποδομή σε όλα τα κράτη-μέλη. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Σας Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αυτές και πραγματικά με βοηθάνε πάρα πολύ να επικεντρωθώ στα σημαντικότερα σημεία της εσωτερικής αγοράς. Σας ευχαριστώ για τα όσα είπατε κυρία Στάιλερ για τις νέες τεχνολογίες, για το ψηφιακό χάσμα. Σαφώς πρόκειται αυτό να μας απασχολήσει και ιδίως το Μάιο θα επικεντρωθούμε στο ζήτημα αυτό. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να προκαταλάβω καθόλου τις αποφάσεις που θα ληφθούν τότε, πάντως σίγουρα τα ζητήματα αυτά θα μας απασχολήσουν και θα δραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην πολιτική μας η διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης. Θεωρείται, έχει αποδειχθεί ότι είναι μια καλή διαδικασία και στην πράξη λειτουργεί. Θέλουμε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία να βασιστούμε. Και είναι πολύ σημαντικό η οδηγία για τις υπηρεσίες να εφαρμοστεί πλήρως σε κάθε χώρα. Ετέθηκε ένα ερώτημα σχετικά με το 10% και τον φόρο επί των εταιριών στην Ουγγαρία. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να επεκταθώ πάρα πολύ στο ζήτημα αυτό και να φερθώ ακόμα και στο παράδειγμα της Ιρλανδίας. Ας μην ξεχνάμε όμως την εποχή εκείνη που ξεκίνησε το 1987 το περίφημο Ιρλανδικό θαύμα. Τότε η Ιρλανδία μείωσε το φόρο της στο 10%, γνώρισε μια τεράστια οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 10% πολλές φορές. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε όμως μια κερδοσκοπική φούσκα η οποία στη συνέχεια έσκασε και προχώρησαν σε διάφορα προβλήματα. Δεν θεωρώ όμως ότι το ποσοστό του 10% συνδέεται άμεσα με τα οικονομικά δεινά της ε, Ιρλανδίας. Για την Ουγγαρία αυτό μπορώ να πω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να στείλουμε το σωστό μήνυμα. Δηλαδή όσοι εργάζονται σκληρά, όσε εταιρείε και όσοι άνθρωποι εργάζονται σκληρά, δεν πρόκειται να τιμωρηθούν. Εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να τιμωρήσουμε αυτού που εργάζονται σκληρά. Για αυτό το λόγο δημιουργήσαμε αυτό τον καταποκοπή φόρο 16% που είναι ο χαμηλότερος στην Ανατολική Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο μειώσαμε τον εταιρικό φόρο από το 19% στο 10%. ιδίω για τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. και πρόκειται να διευρύνουμε την πολιτική αυτή για όλες τις επιχειρήσεις μετά από την 1η Ιανουαρίου του 2013. Το κάνουμε λοιπόν αυτό γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι σε καμία περίπτωση το κράτος δεν θα πρέπει να τιμωρεί τους ανθρώπους εκείνους, επιχειρήσεις εκείνες που εργάζονται σκληρά. Ευχαριστώ. Yeah, that was my first. Anyway. Oh, are you, oh, um, sorry, yes, I missed that. Yeah, okay. Good. Uh, well, Minister, can I... Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρευρεθήκατε εδώ σήμερα το πρωί και απαντήσατε σε τόσες πολλές ερωτήσεις. Και νομίζω ότι θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας στις μελλοντικές μας εργασίες ε, Θέλω να σας πω ότι η Επιτροπή μας θα επισκεφτεί την Ουγγαρία από τις 22 στις 24 ε, Φεβρουαρίου. Ίσως θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε, ίσως σε πιο άτυπο πλαίσιο. Θα είναι πολύ ωραίο να συνεχίσουμε το διάλογο και να περάσουμε και λίγο χρόνο μαζί. Και όπως βλέπετε, οι συναδελφοί μου ενδιαφέρονται πάρα πολύ, όχι μόνο για το έργο σας εδώ, αλλά ε, μας ενδιαφέρει να συζητήσουμε και μαζί σας και με τους συναδέλφους σας στο Υπουργείο Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή τη δέσμευση κυρίως ε, για την πράξη της ενιαίας αγοράς ε, και φυσικά και η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών θα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα έχουμε και σοβαρές συζητήσεις μαζί σας για το πώς θα προωθήσουμε και εκείνο το φάκελο. Αλλά νομίζω ότι συμπερασματικά θέλω να σας ευχηθώ εκ μέρους όλη της Επιτροπής μας ε, κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας γιατί εμείς θεωρούμε ότι η ε, περιτροπής προεδρίας γίνονται όλο ένα και πιο σημαντικές. Έτσι λοιπόν, να ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παραβρεθήκατε εδώ σήμερα το πρωί.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 Uh, κυρίες και κύριοι, ε, θα σας παρακαλούσα να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Παρακαλώ καθίστε. Ελπίζω όλοι να έχετε τις κάρτες ε, σας. Ε, νομίζω... Νομίζω πρέπει να σας έχει ζητηθεί. Άλλωστε έτσι κάνουμε συνήθως στην Επιτροπή μας. Ας ελέγξουμε πρώτα, πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Ας ψηφίσουμε λοιπόν. Θα παρακαλούσα όλα τα μέλη του ΕΛΚ να ψηφίσουν. 11 έχουμε νομίζω. Συγγνώμη Μάλκολμ, έρχεται η κάρτα μου. Η κυρία του μόλις ήρθε. Εντάξει, είσαστε εντός της ποσόστοσής σας. Έρχεται η κάρτα μου. υπολογίστε με και εμένα. Η κυρία Ρόιτοβα, ναι. Η κάρτα σας δεν λειτουργεί. Μπορείτε παρακαλώ να ξαναδοκιμάσετε, διότι δεν ε, ανάβει εδώ το φωτάκι. Ωραία, κλείνω την ψηφοφορία. Ωραία, κατόπιν λαϊκού αιτήματο ε, ξαναψηφίζουμε. Ξαναψηφίζει το ΕΛΚ. Δέκα έχουμε. Κάποιος δεν ψήφισε. Δώδεκα και η κυρία Κανιέτε. Δεκαπέντε συνολικά. Δεκαπέντε συνέσω, δεκατέσσερις. Ωραία. Το ΕΛΚ ε, βρίσκεται εντό τη ποσόστοση του. η ομάδα τη κυρία Κέπχαρτ, SND, ε, οι Σοσιαλδημοκράτε, ε, ανοίγει η ψηφοφορία, αρχίζει η ψηφοφορία. Δέκα, πολύ ωραία. Δέκα για την ομάδα SND. Νομίζω ότι τους άλλους θα τους κάνουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Τρεις φιλελεύθερους βλέπω, τρεις πράσινους. Ε, δύο συνέναν εμένα από το ε, CNR, τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ας προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στην ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας Κέπχαρτ για την εφαρμογή της οδηγίας περιπηρεσιών. Ε, θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Κέπχαρτ να κάνει μια εισαγωγή αν θέλει να πω μόνο ότι θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τους κοιόδης εισηγητές. Ε, χθες το βράδυ ο κύριος Λέκκαρτ και εγώ ε, συμφωνήσαμε. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες κατά την ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. So, let's move on to the vote then. So, um, the... Να προχωρήσουμε λοιπόν. Ε, τροπολογία 12 του κυρίου Καμφέν, Αρχή της ψηφοφορίας. The vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 20 κατά 15 υπέρ. Προχωράμε στην παράγραφο 1β της Επιτροπής Οικονομικών. Ε, χωριστή ψηφοφορία, όπως βλέπετε στο κατάλογο, ζητήθηκε από το ΕΛΚ. Πρώτο μέρος, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος, αρχή της ψηφοφορίας για το δεύτερο μέρος. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 20 κατά, 14 υπέρ. Τροπολογία 13 του κυρίου Καμφάν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 14. Θα πρέπει να ψηφίσουμε τη 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται σαφώς. 15 ε, του κυρίου Καμφάν. Αρχή της ψηφοφορίας για την ε, τροπολογία 15. The vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται 20 κατά 15 υπέρ. 16 των κυρίων Χουάνγκτοκ και Βερνιό. Χωριστή ψηφοφορία ζητήθηκε από την ΕΛΚ. Από, συγγνώμη, από τους φιλελεύθερους. Ε, αρχή της ψηφοφορίας για το πρώτο μέρος. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 20 κατά 16 υπέρ. Το δεύτερο μέρος, ποιος είναι υπέρ, κατά, α, εγκρίνεται. 17 του κυρίου Πουπάκη και της κυρίας Χάνσλι. υπέρ, κατά, εγκρίνεται σαφώς. Τροπολογία 18 ε, του Προέδρου σας, υπέρ, κατά, απόχε εγκρίνεται. Ε, της ε, Επιτροπής Απασχόλησης 2, ε, διότι καταπίπτει διότι υιοθετήθηκε η 18. Η, διο, πάμε στην, στην 12 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά εγκρίνεται σαφώς. Δεν χρειάζεται να μετρήσουμε. Έμπλ 1 υπέρ κατά εγκρίνεται σαφώς. Επιτροπή Αποσχόληση 10, αυτή καλύφθηκε από την 18. Φτάνουμε στην ε, πρώτη της ε, ε, Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης υπέρ, κατά. Εγκρίνεται σαφώ. Η τέταρτη τη Επιτροπής Αποσχόληση. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 15 υπέρ 21 κατά. Εκον 4 καλύφθηκε ήδη. Ε, πάμε στην 3 της Επιτροπής Απασχόλησης. Αρχή της ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορία. Σαφώς απορρίπτεται 22 κατά 15 υπέρ. 15 της Επιτροπής Ρέτζη. Χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος ψηφίζουμε υπέρ, κατά, εγκρίνεται σαφώς. Δεύτερο μέρος, ε, αρχή της ψηφοφορίας για το δεύτερο μέρος. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 20 ε, κατά 17 υπέρ. Ε, πάμε στην 7 της Ρέτζη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σαφώς. Προχωράμε στην Ρέτζη 8 χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο μέρος αρχή της ψηφοφορίας λήξη της ψηφοφορίας Απορρίπτεται. 15 υπέρ, 22 κατά. Νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε το δεύτερο μέρος. Ε, σηκώστε τα χέρια σας. Ποιος είναι υπέρ του δεύτερου μέρους. Κατά. Εγκρίνεται σαφώς. Ρέτζι 9. Αρχή της ψηφοφορίας για την 9 της Ρέτζι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 19 υπέρ 17 κατά. Παράγραφος 20, παράγραφος 4, τροπολογία 20 του κυρίου Μέλτσερ. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 21 του κυρίου Λουκεγκάρντ, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 22 του κυρίου Ότμαρ Κάρας, ε, αρχή της ψηφοφορίας για την τροπολογία 22. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 υπέρ, 16 κατά. Ε, τροπολογία 23 του κυρίου Καράς, υπέρ, κατά. Εγκρίνεται σαφώς. 24 του κυρίου Καμφά, αρχή της ψηφοφορίας για την τροπολογία 24. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η 22 κατά 15 υπέρ. 25 του κυρίου Μέλτσερ. Αρχή της ψηφοφορίας για την 25 του κυρίου Μέλτσερ. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 ε, ψήφοι κατά, 16, ε, υπέρ 16 κατά. 28 ε, του Προέδρου σας. Αρχή της ψηφοφορίας για την τροπολογία 28. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 ψήφοι υπέρ, 16 κατά. 26 της κυρίας Χάνσλικ και άλλων υπέρ, κατά. Εγκρίνεται σαφώς. 27 του κυρίου Λούκεγκαρτ. Ε, προσθήκη. Ε, αρχή της πληροφορίας για την 27. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται 22 υπέρ 13 κατά. 29 του, των κυρίων Χουαγντοκ και Βερνιό υπέρ κατά. Εγκρίνεται σαφώς. 30 του κυρίου Καμφά. ανοίγει η ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας για την τροπολογία 30. Λήξη της πληροφορίας Απορρίπτεται. 22 κατά, 15 υπέρ. Προχωράμε στην 31. Με προφορική τροπολογία ε, την διαγραφή του κεντρικού σημείου της παραγράφου αυτής. 31 ε, του κυρίου Λεκεκάρτ με την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, Εγκρίνεται σαφώς. Η 31 καταπίπτει. 32 του κυρίου Λεγκάρτη υπέρ κατά. Εγκρίνεται σαφώς. 34 του κυρίου Κουπάκη. Αρχή της ψηφοφορίας για την τροπολογία 34. Λήξη. Εγκρίνεται 22 ψήφοι υπέρ, 15 κατά, καταπίπτει 33. Πάμε στην 35 του κυρίου Πουπάκη. Μπορούμε να την ψηφίσουμε υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 36 της κυρίας Κέπχαρτ. Αρχή της ψηφοφορίας για την 36. λήξη της ψηφοφορίας 20 υπέρ 18 κατά 37 του κυρίου Καμφά αρχή της ψηφοφορίας για την 37. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 17 υπέρ 20 κατά. 38 του Προέδρου σας. Αρχή της ψηφοφορίας για την τροπολογία 38. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 25 υπέρ 11 κατά. Προχωράμε τώρα στη συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε, περνάμε τώρα αρκετέ σελίδες και πάμε στην τροπολογία 49 της κυρίας Χάνσλη και άλλων. Τροπολογία 49 υπέρ, κατά, εγκρίνεται σαφώς. 50 της κυρίας Χάνσλη και άλλων υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 51 της ίδιας ομάδας υπέρ κατά εγκρίνεται. Η ΕΚΟΝ 2 ήδη έχει καλυφθεί. Πάμε στην ε, συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά εγκρίνεται σαφώς. Περνάμε στην τροπολογία 58 του κυρίου Πουπάκη υπέρ κατά εγκρίνεται. 59 του Προέδρου σας υπέρ κατά εγκρίνεται. 62 της κυρίας Κέπχαρτ ε, έχει ζητηθεί από το ΕΛΚ χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος υπέρ, κατά εγκρίνεται σαφώς. Αρχή της ψηφοφορίας για το δεύτερο μέρος. Αρχή της ψηφοφορίας για το δεύτερο μέρος της 62. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 23 κατά 14 υπέρ. Προχωράμε στην τροπολογία 60, την κυρία Σεχνάλοβα. Χωριστή ψηφοφορία και πάλι. Ε, το κύριο κείμενο υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και η προσθήκη and the European Parliament υπέρ, ε, συγγνώμη, αρχή της ψηφοφορίας, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται με 21 ψήφους κατά, 17 υπέρ. Τροπολογία 61 της κυρίας Χάνσλικ και άλλων προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται σαφώς. Οι 63 και οι 39 δεν ψηφίζονται διότι εγκρίθηκε η συμβαστική. Πάμε στην 66 του κυρίου Λεκεγκάρτ υπέρ κατά εγκρίνεται. 65 του κυρίου Καφέ υπέρ κατά, εγκρίνεται. 67 του Πρόεδρου σας υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 68 του κυρίου Καμφέ, αρχή της ψηφοφορίας για την 68. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. 22 κατά, 16 υπέρ απορρίπτεται. Προχωράμε στην τροπολογία 69 με προφορική τροπολογία που βρίσκεται στον κατάλογο των, των, της πληροφορίας που έχετε. Ε, υπέρ. Νομίζω μπορούμε να σηκώσουμε χέρια. Ε, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται σαφώς. Η 69 καταπίπτει. 9 της Επιτροπής Αποσχόλησης. Αρχή της ψηφοφορίας για την 9 της Επιτροπής Αποσχόλησης. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 ψήφοι υπέρ, 17 κατά. Παράγραφος 16. Τροπολογία 70 με ε, προφορική τροπολογία υπέρ, κατά. Εγκρίνεται σαφώς. Η 70 καταπίπτει. Περνάω στην 2 της ε, Περιφερειακής Επιτροπής ε, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 4 της Ρέτζη υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ρέτζι 6 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 6 Επιτροπής αποσχόληση υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Να ψηφίσουμε υπέρ, κατά, εγκρίνεται σαφώς. Και προχωράμε τώρα στην ε, τροπολογία 78, παράγραφο 18α νέο, του κύριου Καμφάν. Αρχή της ψηφοφορίας για την 78. Λήξη της ψηφοφορίας. Ε, απορρίπτεται 20 κατά 16 υπέρ. Ρέτζι 10. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 21 ψηφί κατά 16 υπέρ. Ρέτζι 11. Υπέρ κατά, εγκρίνεται σαφώς. Ρέτζι 12, υπέρ, κατά, εγκρίνεται επίσης. 79 του κ. Καμφάν. Αρχή της ψηφοφορίας. The vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 21 κατά 16 υπέρ. Έκον 3 δεν την ψηφίζουμε. 80 ε, του Πρόεδρου σας υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 5 της Επιτροπής Αποσχόλησης. Την ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Open, Αρχή της ψηφοφορίας. Votes closed. That's 23 against 15. Απορρίπτεται 23 κατά 15 υπέρ, 11 της Επιτροπής Απασχόλησης, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται επίσης. Ε, τροπολογία 4 του κ. Καμφά, αρχή της ψηφοφορίας. Ε, Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται επίσης. Η Α της Επιτροπής Απασχόλησης καλύπτεται ήδη από το εκτιμώντας Α, ε, εκτιμώντας Β5 του κ. Καμφά, αρχή της ψηφοφορίας. The Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται επίσης. Έκον α. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Έξι Της κυρίας Λεγκρίπ και άλλων. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Έπτα Του κυρίου Καφέ. Αρχή της ψηφοφορίας. Votes closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 8 του κυρίου Μίλτσερ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται σαφώς. 9 της κυρίας Χάνσλικ και άλλων. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 10 της κυρίας Μπιζότο και άλλων. Υπέρ κατά απορρίπτεται 11 του κυρίου Μέλτσερ υπέρ κατά απορρίπτεται επίσης Β της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά εγκρίνεται η C ήδη έχει καλυφθεί ε, Έκον Β ψηφίζουμε είναι το εκτιμώντας ED, αρχή της ψηφοφορίας για την ΕΚΟΝ Β. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 22 ψήφοι υπέρ 16 κατά. Καταπίπτει η D της Επιτροπής Απασχόλησης, ε, ε της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά εγκρίνεται σαφώς και Τροπολογία 1 του κυρίου Καμφά, αρχή της ψηφοφορίας. Ε, λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 16 υπέρ, 21 ψήφι κατά. 2 του κυρίου Καμφά υπέρ, κατά. Εγκρίνεται σαφώς. Τροπολογία 3 του κυρίου Καμφά υπέρ κατά εγκρίνεται σαφώς. Έτσι ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε το σύνολο της έκθεσης. Αρχή της ψηφοφορίας για το σύνολο της έκθεσης, διότι νομίζω ότι ηλεκτρονικά πρέπει να εγκρίνουμε την έκθεση αυτή. Ψηφίσατε όλοι λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 32 ψήφους υπέρ, μία ψήφο κατά και πέντε αποχές. Ε, θερμά συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας, ε, κυρία Κέπχαρτ. Σας ευχαριστούμε. Um, um, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Και όσοι ήσασταν και εδώ νωρίτερα θα ακούσατε και τον Ούγκρο Υπουργό που αναφέρθηκε στην ε, εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες ε, και είπε την υπομονή για την υιοθέτηση της έκθεσης. Έτσι λοιπόν θα διασφαλίσουμε ότι το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα το συντομότερο θα λάβει ένα αντίγραφο τη έκθεσή μα ε, και ίσω ε, θα μεταβούμε και να τη συζητήσουμε μαζί του. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη μα ψηφοφορία για σήμερα το πρωί. Προχωρούμε τώρα στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης προς ε, επαρκή βιώσιμα και ασφαλή στα συστήματα. Εδώ είναι ο κύριος Ντεγιόνκ, ο εισηγητής. Θέλετε να πείτε δύο λόγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές ε, για την πολύ καλή συνάντηση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο όπου καταλήξαμε σε συμβασμό σε αρκετές ε, συμβαστικές τροπολογίες. Μπορώ να υποστηρίξω και αρκετές προφορικές τροπολογίες ε, που υποβλήθηκαν χθε το βράδυ ακριβώς πριν από την σημερινή συνεδρίαση. Απλώς θέλω να αναφερθώ σε ένα σύνολο τροπολογιών που θα μπορούσε να κάνει λιγότερο ισορροπημένη ε, την ε, έκθεση σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς. Η δυνατότητα μεταφοράς είναι κάτι καλό για να βελτιώσουμε την δυνατότητα κυκλοφορίας, την ελευθερία της κυκλοφορίας των εργαζομένων. Όμως η έκθεση ακολουθεί τη μέθοδο ότι καταρχήν πρέπει να αποτιμήσουμε τα υφιστάμενα προβλήματα και μπορώ να σας διασφαλίσω ότι υπάρχουν κάποια και κατόπιν ε, να δούμε το θέμα της εφαρμογής και ορισμένες τροπολογίες φαίνεται να προτείνω ότι μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στο θέμα της δυνατότητας μεταφοράς και αυτό είναι αντιφατικό κατά κάποιο τρόπο γι' αυτό εγώ τοποθετήθηκα αρνητικά σε κάποιες τροπολογίες ε, κατά τα λοιπά για τις υπόλοιπες ευχαριστώ τους εισηγητές Uh, Ευχαριστούμε πολύ για την εργασία που έχετε κάνει. Ξέρω ότι έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις για να καταλήξετε σε συμβαστικές τροπολογίες. Από ό,τι κατάλαβα έγιναν και κάποιες συζητήσεις την τελευταία στιγμή, ιδίως όσον αφορά τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Εφόσον θα είναι η πρώτη που θα ψηφίσουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω να σας ε, ζητήσω μάλλον, να σας ρωτήσω αν έχετε την τελευταία εκδοχή της συμβαστικής τροπολογίας υπαριθμών 1, γιατί έχει γίνει και πρόταση να γίνει κατά τμήματα εδώ πέρα ψηφορία. Συνήθως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά από ό,τι κατάλαβα το συζητήσετε αυτό με τους σκιώδεις, αν συμφωνούν και αυτοί, τότε και εγώ να ακολουθήσω το αίτημα αυτό. Ήθελα απλώς να εξασφαλίσω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες ε, συμφωνούν με την πρόταση αυτή. Θα μας πείτε λοιπόν τώρα τι γίνεται με τη συμβαστική ναι, ναι, γιατί για τα υπόλοιπα νομίζω τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ όλων των προτάσεων που γίνανε και για την πρόταση για την ξεχωριστή ψηφοφορία. Έχουμε εδώ πέρα μια προφορική τροπολογία από τον κύριο Μάντερς στο τελευταίο τμήμα. Εγώ μπορώ να δεχτώ την προσθήκη αυτή που κάνει ο συνάδελφος. Επί της ουσίας, ουσιαστικά τα πράγματα άλλαξαν κάπως εξαιτία της προφορικής τροπολογίας. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο βασικό περιεχόμενο, πρόεδρος. Λοιπόν, ας είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι έχετε στον κατάλογο ψηφοριών συμβαστικές τροπολογίες. Το πρώτο τμήμα είναι η αρχική παράγραφος 1, 1α και 1β. Στη συνέχεια θα κάνουμε δεύτερη ψηφορία για το 1c, το 1γ Επίσης δέχεστε να ψηφίσετε για την προφορική τροπολογία του κ. Μάντερς, ο οποίος μάλλον θα πρέπει να μας τη διαβάσει κιόλας να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει όλες οι πολιτικές ομάδες να αποδεχθούν την προφορική τροπολογία. Πολύ ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πρώτο τμήμα, 1α και 1β υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στο ένα σ υπέρ, κατά, εγκρίνεται περνάμε στο τρίτο τμήμα, προφορική τροπολογία Manders, που απλώς προσθέθηκε τώρα στην, στον κατάλογο ψηφοριών. Μπορείτε να μας το διαβάσετε. Ναι, σαφώς, Πρόεδρε. Αφού το συμφωνήσαμε με τους σκιώδεις ηγητές, δεν ήταν όμως στον τελικό κατάλογο ψηφοφοριών. Γι' αυτό το λόγο χθε το βράδυ προσπαθήσαμε πάλι να το προσθέσουμε είναι μια προσθήκη στην προφορική τροπολογία που λέει ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης θα προσπαθήσουν μαζί να εκπληρώσουν τις ταξιδιωτικές υποχρεώσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν ε, διασυνοριακή επίπτωση. Κάλυψη δηλαδή των ε, στεξιωτικών υποχρεώσεων και διασυνοριακά. Δεν νομίζω ότι αντιτίθεται κανεί σε αυτό, επομένω ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για το τελευταίο αυτό τμήμα. Πέρας. Ναι, ναι, τη δική σας τροπολογία ψηφίζουμε. Ναι, έχει εγκριθεί το άλλο. Ναι, έχει εγκριθεί. Πρέπει να έχετε ψηφίσει ουσιαστικά. Εγκρίνεται λοιπόν και επίσημα. Περνάμε τώρα στις υπόλοιπες τροπολογίες. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, γιατί ξαφνικά τώρα έχω δύο έντυπα μπροστά μου. Περνάμε στην τροπολογία 6. Υπέρ. Μάλλον ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 6. One Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 23 υπέρ 14 κατά. 8 του κύριου Γκρέκ. άρθη ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Είστε όλοι υπέρ, δεν χρειάζεται τότε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 της κυρίας Τούρνεν. Υπέρ. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρο. ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε για την τροπολογία 7 τη κυρία Τούρουνεν. Άρτη ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. 13 υπέρ, 24 κατά. Τροπολογία 9 του κυρίου Λουί Γκρέκ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 του κυρίου Έγγελ. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 23 υπέρ, 15 κατά. 12 του κυρίου Ζουβάν και Έγγελ. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 13 Λουίς Κρέκα έχει αποσυρθεί, 14 Ζουβάν και Έγγελ. Υπέρ. Κατά. Α το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά, λέει ο πρόεδρο. Τροπολογία 14. Άρτη ψηφοφορία. Έχει εγκριθεί. Τροπολογία 15 του κ. Χουαγνόγκα. Άρτη ψηφοφορία για την τροπολογία 15. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 17 της κυρίας Τούρουνεν. Άρχεται ψηφοφορία για την τροπολογία 17. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20 Λουί Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 21 του Ρούνεν. Άρτε ψηφοφορία για την τροπολογία 21. Πέρας. Απορρίπτεται 18 υπέρ 20 κατά. Τροπολογία 22 της κυρίας Τούρουνεν. Άρχεται ψηφοφορία για την τροπολογία 22. Πέρας. Εγκρίνεται 22 υπέρ 16 κατά. Τροπολογία 23 Κρόιτσμαν. Άρχεται ψηφοφορία για την 23. Πέρας. Εγκρίνεται 22 υπέρ 15 κατά. Τροπολογία 24 του κυρίου Κρότσμαν πάλι. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία και πάλι. Τροπολογία 24 του κ. Κρότσμαν, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται ξεκάθαρα. 8 υπέρ 20 κατά. 9 αποχές. 25 του κ. Μόλτσερ. Άρτε ψηφοφορία για την τροπολογία 25. Πέρας. Απορρίπτεται. 26 της κυρίας Τούρουνεν. Άρχεται ψηφο... Μάλλον, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται ξεκάθαρα. Τροπολογία 27 του κύριου Γκρέχ. Που είναι προτείνω να διαγραφούν οι λέξεις ε, μέσω του εισαγωγής του δεύτερου και τρίτου πυλώνα, να μπει το συμπλεκτικό end και, και θα έχουμε το ακόλουθο. Καλή τα κράτη-μέλη που δεν έχουν υποβάλει συγκεκριμένα σχέδια, που, ξεκάθ, που έχουν ξεκάθαρα και ποσοτικοποιημένους στόχους, για την ε, διαμόρφωση των στεξιωτικών συστημάτων να ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό το στομότερο δυνατό προκειμένου να επιτρέψουν στους καταναλωτές και τους πολίτες να γνωρίζουν ακριβώς πώς θα διαμορφωθεί η μελλοντική του σύνταξη. Δεν είμαι σίγουρος ότι χρειάζεται το συμπλεκτικό και, λέει ο Πρόεδρος, στα αγγλικά τουλάχιστον. Νομίζω ότι μπορούμε και στη συνέχεια να το διευθετήσουμε γλωσσικά. Ποιοι είναι υπέρ τις τροπολογίες όπως τροποποιήθηκε. Κατά εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 3 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Περνάμε στη τροπολογία 32 του κυρίου Πουπάκη. Άρτη ψηφοφορία για την 32. Πέρας εγκρίνεται 21 υπέρ 15 κατά. Συμβαστική τροπολογία 4 του εισηγητή και άλλων υπέρ κατά εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 36 της κυρίας Τούρουνεν. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 38 του κυρίου Μάντερς. Άρτη ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 38. πέρας. Εγκρίνεται 21 υπέρ 15 κατά. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία Ψηφίζουμε για το σύνολο της γνωμοδότησης ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται ξεκάθαρα 34 υπέρ, 3 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια στον κύριο Ντιγιόγκ. Σας ευχαριστούμε πολύ. και ελπίζουμε ότι θα υπερασπιστείτε τη γνωμοδότησή σα στην Επιτροπή Απασχόληση. Περιμένουμε νέε επιτυχίε εκεί πέρα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ όλου για την ψηφοφορία. Θα κάνουμε ο ολιγόλεπτο διάλειμμα και συνέχεια θα συνεχίσουμε με την συνεδρίαση των συντονιστών στι 11 παρατέταρτο. Η επόμενη συνεδρίαση τη Επιτροπή μα θα γίνει την 3η 1η Φεβρουαρίου. 9 με 6.30 και αν όλα πάνε καλά θα ψηφίσουμε για την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Αυτή λοιπόν θα είναι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Λύεται συνεδρίαση.